Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη της κοινή συνεδρίασης ε, με θέμα την δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Χθες είχαμε μία ανευπροηγουμένου εκδήλωση και συνεδρίαση. Είχαμε ακρόση με 7 πρωθυπουργού, ε, με 7 συγγνώμη, υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Και διαπιστώσαμε από την ανταλλαγή απόψε που είχαμε χθε ότι δεν υπήρχε απόλυτη σύγκληση απόψεων. Αλλά είναι σημαντικό και οι υπουργοί να έρθουν σε επαφή με το Κοινοβούλιο. Και για αυτού είναι σημαντικό, αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σημαντικό να έχει άμεση επαφή με αυτού που σχηματίζουν τι κυβερνήσει και όχι με ε, τον εκπρόσωπο απλώ τη Προεδρία που αλλάζει κάθε εξάμεινο. Πραγματικά δεν είχαμε τέτοια ευκαιρία προηγουμένως. Ήταν πρωτοφανής και ελπίζω να επαναληφθεί. Θα ακούσουμε τώρα τους συνεισηγητές. Έχουν λάβει πληθώρα τροπολογιών και θα μας εξηγήσουν αν ήδη έχουν αρχίσει να σκεγγραφούνται κάποιες συμβαστικές τροπολογίες. Δεν ξέρω ποιος θα δώσει τον Αρκτήριο λάκτισμα της συζήτησης. Ο Έρμαρτ Μπέγκεφ ίσως. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που δεν μπορούσα να είμαι εδώ χθε το βράδυ, γιατί στην περιφέρειά μου γινόταν ο ε, διορισμός για, τους, ε, για τον, για τον υποψήφιο τους υποψηφίους για τις εκλογές ε, της επόμενης χρονιάς. Δυστυχώς δεν μπορούσα να είμαι λοιπόν παρόν. Παρόλα αυτά, ε, χαίρομαι πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, είναι βεβαίως πάρα πολύ νωρίς για να παρουσιάσουμε ένα πακέτο συμβιβαστικών τροπολογιών, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά. Έχουμε προβλέψει ένα χρονοδιάγραμμα, ώστε πριν από τις, ε, πριν από τις 29... Ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι, θα εργαστούμε ε, πολύ εντατικά την επόμενη εβδομάδα. Ε. Έχουμε μία ε, συνεδρίαση με τους σκιώδεις εισηγητές για τις παραγράφους 1 έως 16. Ήταν πάρα πολύ επικοδομητική η συνεδρίαση αυτή και μετά από αυτήν ε, θα προχωρήσουμε στα, επόμενα, στα υπόλοιπα σημαντικά ζητήματα. Να σας αναφέρω κάποια στοιχεία τα οποία μου φαίνονται χρήσιμα και είναι σημαντικό να υπάρξει μία απάντηση για τα 1 ως 16 υπάρχει ένα ερώτημα όσον αφορά την, ε, το, το, την εφαρμογή του Συμφώνου ε, Σταθερότητας, τι θα κάνουμε, επειδή πολλές φορές τα κράτη-μέλη δεν, δεν σέβονται το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Δεύτερον, το ρόλο των ειδικών αναχώρασης τάσεων, ε, πώς θα μπορούσαμε να τους να βοηθήσουμε. Ε, και τον ε, κώδικα που ήδη ε, ψηφίστηκε και εγκρίθηκε. Αυτό είναι επίσης ένα θετικό στοιχείο. Και τρίτον, ένας μηχανισμός απορρόφησης των κρίσεων. Και από αυτού πρέπει να συζητήσουμε διεξοδικότερα, γιατί ένα είναι σαφές, εμείς ως εισηγητές παρουσιάζουμε δύο επιλογές. Υπάρχει μία συζήτηση αυτή τη στιγμή, ένα εργαστήριο που θα γίνει μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές και σας υπενθυμίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε μία έκθεση με ε, σκέψεις για, ε, για το πώς θα μπορούσε να είναι ένας τέτοιος μηχανισμός απορρόφησης κρίσεων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, γιατί έχουμε τροπολογίες που πηγαίνουν προς τρεις διαφορετικές ε, κατευθύνσεις και θα πρέπει να επιλέξουμε να βρεθεί μια πραγματική ισορροπία, κάτι το ρεαλιστικό. Και όταν λέω ρεαλιστικό, εγώ εννοώ ένα ρεαλιστικό όραμα, ε, καλά ε, μέσα, ε, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2001 ήδη και το 2003 ε, ήδη πρότεινε την ακτοφυλακή την ευρωπαϊκή και τώρα έχουμε αρχίσει να προσπαθούμε να ε, την ιδρύσουμε. Είναι λοιπόν πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε εκ των προτέρων συζητήσεις, να είμαστε έγκαιροι για να μπορέσουμε να ε, προβούμε σε πρόληψη και να σταθεροποιήσουμε την Ευρωζώνη. Υπάρχει το θέμα των δημοσιονομικών πτυχών και το θέμα των ιδίων πόρων. Βεβαίως περιμένουμε και τη ε, επί των ιδίων πόρων που θα λάβει η χώρα το Σεπτέμβρη και υπάρχουν και διάφορες τροπολογίες ε, που αφορούν το πώς ε, θα εμπλακούν τα εθνικά κοινοβούλια, πώς θα γίνει να μην μπούμε στα χωράφια των εθνικών κοινοβουλίων και να δούμε τις σχετικές αποφάσεις του δικαστηρίου, τι θα κάνουμε με τις ε, συνθήκες κλπ. κλπ. Όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα εμβαθύνουμε περισσότερο και οι συζητήσεις αυτές πρέπει να είναι δημόσιες. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, το είδος των μέσων, ο ρόλος των μηχανισμών σταθεροποίησης, ε, ποιος πρέπει να είναι, ποια πρέπει να είναι η σχέση με ε, το Διεθνές Νομισματικό ε, Ταμείο, μηχανισμός λοιπόν σταθερότητας και πώς μπορούμε να χωρίς να αλλάξουμε τις, τις συνθήκες, να προχωρήσουμε, να μην χάσουμε χρόνο και να προετοιμάσουμε τη δεύτερη φάση, να κάνουμε κάποιες αλλαγές στις συνθήκες για να δούμε πού θέλουμε να φτάσουμε, ποιος είναι ο τελικός μας προορισμός. Εκεί πρέπει να είμαστε βέβαια προσεκτικοί. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις επιτροπές ΑΦΚΟ, με τον κύριο Μπροκ ε, και τον κύριο Φερχόφστα του ή άλλως είμαστε σε επαφή με τους συζητητέ, ε, ώστε να αποφύγουμε τις αποκλήσεις. Δεν θα ήταν καλό αυτό για κανέναν. Και τέλος, το ερώτημα του χάρτη πορείας. Εδώ χρειαζόμαστε προσανατολισμούς από πλευράς πολιτικών ομάδων για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε ο ε, συμβιβασμός μας να γίνει αποδεκτός από όλους. Η κυρία Μπερέζ. Ευχαριστώ. Η συλλογική ευφία που αναπτύσσουμε με τον ε, κύριο Μπέγκε με καθιστά σχεδόν περιττή στην, ε, σε ό,τι αφορά μια εκτενή παρουσίαση. Θα περιοριστώ σε λίγα σχόλια. Σε ό,τι αφορά την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και σας παραπέμπω και σας παροτρύνω να ρίξετε μια ματιά. Όχι γιατί λέει τα ίδια πράγματα, δεν θυμίζουμε γι' αυτό, αλλά πραγματικά και η μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου παρουσιάζει με όλο το γνωστό κύρος αυτού του οργάνου που είναι αναπόφευκτο και για την πρόοδο και της οικονομικής διακυβέρνησης της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης ε, σε αυτά τα θέματα, δίνει τη βάση ε, και τη σωστή τεκμηρίωση και της δικής μας ε, θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμφωνώ με το συμπέρασμα του κύριου Μπέγκε σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Είναι ένα θέμα που αρχίσαμε να το συζητάμε πριν από πάρα πολύ καιρό. Και στη χθεσινή συζήτηση που είχαμε με τους Υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, ε, μια πραγματικά εντυπωσιακή εκδήλωση και πρεμιέρα άνευ προηγουμένου. Εκεί είχαμε κάποιες ε, τριβές. Μετά το Brexit, μετά το δημοψήφισμα του Brexit, εκδηλώθηκαν ανησυχίες για τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια υπερβολικά μεγάλη επιτάχυνση ε, τη συζήτηση του θέματος ε, του προϋπολογισμού της Ευρωζώνης. Οι δύο συνεισηγητές όμως κρίνουν ότι δεν πρόκειται να εξέλθουν σε την προσέγγιση του προϋπολογισμού της Ευρωζώνης ε, με αμυγός θεσμική προσέγγιση. Γι' αυτό και στην τροπολογία 12 έχουμε μια τροπολογία στην οποία διατρανώνουμε και πάλι την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της συζήτησης στο γενικότερο πλαίσιο των προκλήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καμία περίπτωση θέλουμε μόνο θεσμική προσέγγιση. Γιατί τέτοιου είδους απλώς θεσμική προσέγγιση δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών. Απλώς δίνει την εντύπωση ενός ζώου που κυνηγάει την ουρά του. Κάτι άλλο με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, όπως είπε ο Ράιμερ Μπέγκε, κάναμε έναν επιμερισμό των, του έργου και είπαμε ότι τα θέματα διακυβέρνησης ε, θα έχουν ε, περίπτωση θέση στις εκθέσεις της ΑΦΚΟ και αυτοί θα έχουν το πιδάλιο της κατάστασης ε, και σε ό,τι αφορά το ποσοστό του κώδικα σύγκλησης και του τρόπου χρηματοδότησης, εμείς, οι δύο επιτροπές ΕΚΟΝ και Budget, θα πρωτοστατήσουμε. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων σε τρία σημεία. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την ενοποιημένη έκθεση που σας μοιράσαμε. Για την ενοποιημένη αυτή έκθεση δεν έχουμε καταθέσει εμείς ε, δικές μας τροπολογίες, αλλά τροπολογίες που έχουν συνυπογράψει και άλλοι συνάδελφοι και έχουμε αναθεωρήσει την αρχική εκδοχή συμπεριλαμβάνοντας και τις τροπολογίες των συνεισηγητών. Κάτι που δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, απλώς σας δίνει μια ιδέα για το πώς ε, προχώρησε, προχώρησε, προχώρησαν οι σκέψεις μας από την έναρξη των εργασιών μέχρι σήμερα. Θα ήθελα εντάχει να σταθώ σε τρία θέματα που θα χρειαστεί να διορθώσουμε κάπως, να τροποποιήσουμε. Αν δεν κάνω λάθος έχουν κατατεθεί 836 τροπολογίες ε, και σε αυτές θα χτίσουμε κάποιες χρήσιμες συμβαστικές τροπολογίες. Καταρχήν, σχέση μεταξύ χωρών εντός της Ευρωζώνης με τις χώρες εκτός της Ευρωζώνης. Ήταν από την αρχή μία από τις βασικές μας ε, ανησυχίες. Γιατί ακόμη και μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου, σκεφτόμασταν ότι ίσως μετά τις 23 Ιουνίου θα πρέπει περισσότερο να ασχοληθούμε με την Ευρωζώνη ή να μην ασχοληθούμε με ένα θέμα που διχάζει περαιτέρω την Ευρώπη. Εμείς αντίθετα πιστεύουμε ότι ειδικά μετά τις 23 Ιουνίου θα πρέπει να μιλήσουμε για την Ευρωζώνη, αλλά να την παρουσιάσουμε ως μια ζώνη χωρίς αποκλεισμούς και στην οποία όλοι προσβλέπουν κάποια στιγμή να ενταχθούν. Ένα άλλο θέμα. Τρόπος χρηματοδότησης και συνδυασμός ή ε, σχέση προϋπολογισμού της Ευρωζώνης με τον ενωσιακό προϋπολογισμό. Οι σοσιαλιστές, αν δεν κάνω λάθος, κατέθεσαν την τροπολογία περιθμό 425. Σας ε, παρατρύνω να τη διαβάσετε γιατί σου αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω διαμόρφωση τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα θέμα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Και τρίτο τελευταίο σημείο, η συζήτηση για το δημόσιο χρέο. Ακόμη και στην δική μου πολιτική οικογένεια ανέκυψε το θέμα αυτό μέσω κάποιων τροπολογιών. Η τροπολογία 441, κατά τη γνώμη μου, θα μας ε, επιτρέψει να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ των διστάμενων απόψεων, χωρίς να χρειαστεί να αφισβητήσουμε σημαντικές θέσεις μας. Να, ναι. να δώσουμε τώρα τους, ε, το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Προτείνω τέσσερα λεπτά το πολύ για να μπορέσουν όλοι να λάβουν το λόγο και μετά θα κάνουμε και catch the eye. Λοιπόν, και μετά τότε θα είναι δύο λεπτά ε, για τον κάθε ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και του εισηγητέ για τα σχέδια των εκθέσεων, αλλά και για τη δουλειά που έκαναν στι πολλαπλέ συναντήσει και οδών, τι οποίε είχαμε ω τώρα, και όλε του πραγματικά ήταν εξαιρετικά επικοδομητικέ. Το βασικό ερώτημα το βασικό θέμα από το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε όταν μιλάμε για τη δημοσιονομική ικανότητα είναι το τι χρειάζεται η οικονομία μας, τι μπορούμε να πετύχουμε μέσω της δημοσιονομικής μας ικανότητας για να καταστήσουμε την οικονομία μας πιο ανθεκτική ε, σε ό,τι αφορά και τις ενδεχόμενες μελλοντικέ κρίσεις. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε, θεωρώ, από τα αίτια της προηγούμενη προηγούμενης κρίσης. Έλλειψη ανταγωνιστικότητας, ένα πολύ ευάλωτο τραπεζικό σύστημα, και γίνεται φυσικά ε, σημαντική δουλειά σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση και την διακυβέρνηση του, του οικονομικού χώρου. Υπάρχουν λοιπόν ε, Κανόνε δεν υλοποιούνται όμω, δεν εφαρμόζονται. Χρειαζόμαστε πιο πολλού, δεν πιστεύω. Χρειαζόμαστε πιο ευέλικτου κανόνε και πάλι πιστεύω πω όχι. Θα πρέπει να βρούμε το πώ θα μπορούν με ασφαλή τρόπο να εφαρμοστούν αυτές, αυτοί οι κανονισμοί. Τα πράγματα είναι παγωτεύτα Ξέρουμε ότι οι χώρε χρειάζονται μεταρρυθμίσει και οι οποίε και περιλαμβάνονται στι συστάσεις αναχώρα δεν υλοποιούνται όμω. Έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση χθε με του υπουργού και υπάρχουν δύο σκέλη στη συζήτηση. Υπάρχουν μεταρρυθμίσει που δεν κοστίζουν χρήματα. Αυτέ θα πρέπει να γίνουν σε εθνικό επίπεδο. Και δεν κατανοούμε και από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν δεν υλοποιούνται αυτέ οι μεταρρυθμίσει. Υπάρχουν ύστερα μεταρρυθμίσει οι οποίε κοστίζουν χρήματα και θα πρέπει, θεωρώ, να υποστηρίζονται από την δημοσιονομική ικανότητα και θα πρέπει να κάνουμε διάκριση του τι μπορεί να γίνει βράχη πρόθεσμα χωρί συνταγματική τροποποίηση, τροποποίηση των συνθήκων και σε αυτά να επικεντρωθούμε για να υπάρξει και κάποια προστιθέμενη αξία. Και να συζητήσουμε και για τα πιο φιλόδοξα μακροπρόθεσμα βήματα, τα οποία στη τελική ανάλυση θα χρειαστούν κάποια ε, τροποποίηση των συνθηκών. Κάτι άλλο το οποίο ακροθυγώς μόνο το θίξαμε χθε. Ε, το θέμα της ε, χρηματοδότηση της δημοσιονομικής ικανότητας. θα πρέπει να δούμε καταρχά ε, τι χρήματα έχουμε στη διάθεσή μα και από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα το οποίο θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Και δυστυχώ οι, απο... οι απαντήσει των υπουργών χθε ήταν μάλλον απογοητευτικέ. θα και μία ακρόαση με εμπειρογνώμονα στο τέλη Αυγούστου για θέματα τέτοια ε, ταμείων. Θα πρέπει να αποφύγουμε τον ηθικό κίνδυνο των διαρκών ε, μεταφορών χρημάτων και θα θέσουμε και θέματα ρεσιμότητα. Αυτά θα τα δούμε στην ακρόαση τέλη Αυγούστου σε ό,τι αφορά την ανεργία και το μηχανισμό απασχόλησης. Ε, οι συνάδελφοι από το από την ΕΚΟΝ ήταν αντίθετη και γιατί δεν πιστεύουμε ότι το σχέδιο εγγύησης για τους ανέργους είναι εφικτό. Πιστεύουμε ότι σε εθνικό επίπεδο συνδέεται πάρα πολύ στενά με τα σχέδια συνταξιοδότησης, τα οποία διαφέρουν ιδιαίτερα από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Σε ό,τι αφορά τα, τις ε, εισφορές, σε ό,τι αφορά τις τα ποσά που δίδονται, όλα αυτά μας τα εξήγησε η κ. Τέσσελ Μπλουμ χθες. Ε, υπάρχουν λοιπόν και πολιτικής σε πολλές ε, σοβαρές συνέπειες. Ήταν δύσκολο να εξηγήσουμε στον κόσμο εν το μέσο της κρίσης ότι θα χρειαστεί να πληρώσει για τους ανέργους μιας άλλης χώρας, κράτους μέλους. Ε, και μάλιστα σε μια τέτοια κρίση συμμετρική, όχι ασύμμετρη, όπου όλοι είναι δύσκολο λοιπόν να εξηγήσουμε στο λαό μια χώρα ότι θα πρέπει να υποστηρίξει του ανέργου σε μια άλλη χώρα. Και κλείνοντα, υποστηρίζω απόλυτα αυτά που είπαν οι συγητέ. Νομίζω ότι η κυρία Περβάν Σπερέσα αναφέρθηκε ενδελεχώ στην δυνατότητα των χωρών εκτό Ευρωζώνη να συμμετέχουν στο δημοσιονομικό, στη δημοσιονομική ικανότητα. και στην προετοιμασία, στη φάση προετοιμασία ε, ένταξη στην Ευρωζώνη, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα ε, συμμετοχή στη δημοσιονομική ικανότητα. Αν αυτό θα βοηθήσει τι οικονομίε του να γίνουν πιο ανταγωνιστικέ, θα βοηθήσει και την Ευρωζώνη και θα του προετοιμάσει και από πλευρά διακυβέρνηση. Πολύ σα ευχαριστώ και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Σα ευχαριστώ κύριο Τάν. Ευχαριστώ πρόεδρε και χαίρομαι που υπάρχει αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Έγινε και μια συζήτηση στις συναντήσεις των σκιωδών, αλλά είναι καλό που γίνεται και δημόσια αυτή η συζήτηση. Νομίζω ότι πραγματικά το εγχείρημα αυτό, η άσκηση αυτή, είναι κρίσιμη σημασία προκειμένου να τραπηθεί η Ευρωζώνη. Αλλά για να υπάρχει και σαφήνεια για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Πέραν τούτου, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές στην προσέγγιση μας. Και το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε χαρτογράφητα ύδατα δυσκολεύει το όλο εγχείρημα, αλλά πραγματικά αυτό αποτελεί και την ουσία της έκθεσης. Άρα τι αναζητώ. Μία σαφή κατανομή των ευθυνών. Ποιο κάνει τι. Αυτό θεωρώ ότι είναι ουσιοδό σημασία σε, σε όλη τη φάση τη ε, διαδικασία. Έχουμε τις εθνικές πολιτικές, έχουμε και την ε, ε, δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Και αυτό με οδηγεί στο επόμενο θέμα, στο επόμενο ερώτημα. Ε, πώς κατατάσσονται και σε τι σχέση βρίσκονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι κρίσιμη σημασία σε αυτά. Και η διακυβέρνηση είναι θέμα κρίσιμο. Οι κανόνες, ακούσαμε, δεν τηρούνται πάντα. Και ο λόγος είναι ότι τα Εθνικά Κοινοβούλια, οι Εθνικές Κυβερνήσεις, δεν ε, έχουν την αίσθηση ότι πρόκειται για δικέ του πολιτικέ, για δικού του κανόνε. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στι εθνικέ δομέ να υπάρχει η αίσθηση τη ιδιοκτησία των ε, ε, κανονισμών αυτών. Επίση, έχουμε τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό, την Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική Ικανότητα και είναι σημαντικά τα σκέλη αυτά και για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό αλλά και για το Δημοκρατικό Έλεγχο. Και πραγματικά και εγώ ελπίζω η 425 τροπολογία να μας βοηθήσει να συνδυάσουμε τα δύο σκέλη αυτά κατά κάποιο τρόπο. Γιατί θεωρώ ότι εδώ θα χρειαστούμε μια σαφή απάντηση στο τέλος της έκθεσης. Πολλά θα πρέπει να διευκρινιστούν επίση σε σχέση με τον προπολογισμό μεταξύ άλλων με το θέμα των ιδίων πόρων του Κοινοβουλίου, το οποίο σχετίζεται το δίχως άλλος με την πολιτική αστάθεια που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι αναγκαίο κακό. Αλλά βλέπουμε επίσης ότι εντακτικοποιούνται οι δραστικές μεταρρυθμίσεις και αυτό φυσικά συνδέεται με τη δημοσιονομική ικανότητα, αλλά αποτελεί και μια γενικότερη, ευρύτερη ιδέα πέρα από τα όρια της δημοσιονομικής ικανότητας. Τέλος, για την σύγκληση χρειαζόμαστε επενδύσει και πραγματικά υπάρχει έλλειμμα επενδύσεων στην Ευρώπη στην παρούσα ε, θετία. Ιδρύθηκε το Ταμείο Γιούγκερ, αν και μόλις διάβασα σήμερα ότι απαγορεύεται να τη χρησιμοποιώ αυτό ως όρο. Αλλά πρόκειται για ένα μέσο. Αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά στην Ευρώπη είναι επενδύσεις, γιατί μόνο έτσι θα πετύχουμε σύγκληση μέσω ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προβλέπετε κάπου και στον ευρωπαϊκό προπολογισμό το θέμα των επενδύσεων και προσβλέπω στι περαιτέρω συζητήσει. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Κιόλ. Ο οποίο όμω δεν είναι στην αίθουσα. Δεν είναι πια εδώ ο κύριο Κόλμελ. Η κυρία Πύρκο είναι κάπου εδώ. Ευχαριστώ, Και να ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση. Δεν μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ιδέα ότι η δημιουργία ε, ενός Ευρωπαϊκού Υπουργείου Οικονομικών προβάλλεται ως λύση γιατί αυτό αποτελεί ένα κλασικό, μια κλασική απάντηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόβλημα με την οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη, ωστόσο, δεν είναι η έλλειψη θεσμικών οργάνων, αλλά η έλλειψη εφαρμογή κανόνων. Το πιο προφανέ παράδειγμα είναι ο κανόνας για το δημοσιονομικό έλλειμμα, το οποίο δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 3% σε σχέση με το ΑΕΠ. και έτσι ό,τι αφορά το δημοσιοχρέο στο όριο του 60%. Αυτό προβλεπόταν ήδη από τη συνθήκη του Μάστριχτ. Και έθεσε τη βάση για το ευρώ. Δεν χρειάζεται να σας πω ποιε είναι οι χώρε που το παραβίασαν. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν χώρε που να μην το έχουν παραβιάσει κιόλα. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Η δική μου τροπολογία προτείνει να προσεγγίσουμε εκ νέου το πνεύμα της συνθήκης του Μάστραχτ. Σαφής και υλοποιήσιμες κυρώσεις εις βάρος των κρατών μελών που δεν τηρούν τους κανόνας. Τούτου του λεχθέντους. Κάποιες χώρες δεν ε, πρέπει να εξαναγκάζονται να παραμείνουν στην Ευρωζώνη κατά τη θέλησή τους. Γι' αυτό λοιπόν κατέβαλα, υπέβαλα και μία τροπολογία η οποία διευκρινίζει ότι αν υπάρχουν χώρες που θέλουν να φύγουν από την Ευρωζώνη θα πρέπει να την έχουν αυτή την δυνατότητα υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕΠ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. De me donner la parole. Θα μου δώσω το λόγο αν μου επιτρέπετε. Είμαι σκιώδης για την ομάδα των φιλελευθέρων. Νομίζω ότι η Ευρωζώνη είναι κάτι πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να στοχεύουν στο να έλθουν στην Ευρωζώνη. Σε επίπεδο μεθοδολογικό υπάρχουν κάποια προήμια θέλουν από αυτή της μεθόδου που ακολουθούμε. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι βέβαια ότι κάθε μία από τις χώρες καταθέτει τους προϋπολογισμούς της, ε, ε, την, ε, τις εγγυήσεις τις οποίες δίδει με ομοιογενή βάση. Οπότε μένει πολλά να γίνουν ακόμα έτσι ώστε οι παρουσιάσεις των οικονομιών των κρατών μελών να είναι αναγνώσιμες. Προς το παρόν αυτό γίνεται με πολύ διαφορετικό τρόπο και είναι δύσκολο να συγκρίνει κανείς και ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται η συμμετοχή στον προϋπολογισμό της μιας χώρας, κάθε χώρας, ε, διαφέρει. Θα πρέπει να εμείνουμε επίσης λοιπόν σε αυτόν τον κώδικα σύγκλησης. Αυτός ο κώδικα σύγκλησης α, φυσικά προαπαιτεί να υπάρχει μια ευελιξία. Δεν θα πρέπει εμείς ε, να βάλουμε ε, στενά ρούχα τις χώρες. <clears throat> θα πρέπει όμως να έχουμε πλαίσια στο εσωτερικό των οποίων οι εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να συγκλίνουν. Σχετικά με την παραγωγικότητα τώρα και το κόστος της εργασίας, σχετικά με τις συντάξεις, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση σε κάθε χώρα και θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο στο μέγιστο δυνατό βαθμό να φέρουμε κοντά τις διακανονιστικές ρυθμίσεις η κινητικότητα των εργαζομένων, όπως επίσης και η κοινωνική προστασία της οποίας θα πρέπει να χαίρουν, ε, είναι ένα σημείο στο οποίο απαιτείται περισσότερη σύγκληση. Στον δημοσιονομικό τομέα έχει υπάρξει πρόοδος ε, για το ποσοστό επιβολής, σαν παράδειγμα στα κέρδη των επιχειρήσεων. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλοί οι οικονομικοί εταίροι χρησιμοποιούν τις ε, ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις, το κάνουν αυτό γιατί οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλαπλασιάζουν τα ειδικά καθεστώτα εξε, εξαίρεσης, τα rulings, τα tax rulings, είναι στην ουσία ανταγωνισμός ανάμεσα στις χώρες που δίδει χώρο ε, στην ε, μορφή αυτή εξαιρέσεων. Είναι μια πρακτική η οποία δεν θα πρέπει να συνεχιστεί. Το ίδιο ισχύει επίσης και για τους τρόπους χρηματοδότησης της κοινωνικής πρόνοιας. Θα συνεχίσουμε την χρηματοδότηση της πρόνοιας αυτής φορολογώντας την ίδια την εργασία. Ή μήπω θα πρέπει περισσότερο να στραφούμε σε μια μεγαλύτερη φορολογία της κατανάλωσης. Η φορολογία στην εργασία είναι φορολογία στην παραγωγή και οδηγεί μεθοδικά στην αύξηση της ανεργίας. Έρευνα και ανάπτυξη. Και εδώ υπάρχει μια μορφή αλληλεγγύης που θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Το ίδιο ισχύει και για τις επενδύσεις και υποδομές. Να επιμείνουμε επίσης στην ανάγκη εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων. Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε εδώ από το Κοινωνικό και Οικονομικό Συμβούλιο να δημιουργήσει μια ομάδα ευρωζώνης στο εσωτερικό της, και έτσι οι σκέψεις που γίνονται σε σχέση με την Ευρωζώνη να μην είναι αυστηρά οικονομικές και να έχουν και μια κοινωνική διάσταση και να μπορούν έτσι οι κοινωνικοί εταίροι στο εσωτερικό της Ευρωζώνης να ανταλλάσσουν τις προσδοκίες τους, τις επιφυλάξεις τους και τις ανησυχίες τους. Έτσι λοιπόν θα μπορέσουμε εμείς ε, να αξιολογήσουμε σωστά τις αρετές της ζώνης ευρώ. Ο κύριος Τόρβαλτς, αν δεν είναι εδώ, η κυρία Νι Ρίαντα. Όχι, ο κύριος Δεμάζη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους συζητητές για τη δουλειά που έχουν κάνει. Καταρχήν, θα ήθελα ε, να πω ότι ε, Πιστεύω ακράδαντα ότι έχουμε και θα έχουμε ασύμετρους κραδασμούς στην Ευρωζώνη. Το είδαμε από την αρχή της κρίσης και έχουμε διαφορετικά επίπεδα πληθωρισμού, ποσοστά πληθωρισμού στα κράτη-μέλη, έχουμε διαφορετικά επιτόκια στα κράτη-μέλη και ταυτόχρονα προσπαθούμε να έχουμε μια σύγκληση των τιμών. Αλλά δεν θα έχουμε ούτε τον μακροοικονομική σταθεροποίηση των νοτίων χωρών. Βέβαια, μια επιπόλη ανάλυση ε, επικρίνει την Ευρωζώνη και το υψηλό δημόσιο χρέος. Αλλά το είδαμε και στην Ισπανία και στην Ιρλανδία ότι ε, το ιδιωτικό χρέος επίσης είναι πολύ σημαντικό και θέλουμε να ε, κάνουμε πιο αυστηρές δημοσιονομικές πολιτικές. Το θέμα είναι ποιος αναλαμβάνει την ισορροπία. Γιατί και τα κρατημέρια θα πρέπει να μειώσουν το δημόσιο χρέος. Αλλά τι σημαίνει αυτό ότι οι επιχειρήσεις και τα η νοικοκυριά θα πρέπει να αυξήσουν το ιδιωτικό του χρέο, γιατί αυτό είναι ο βασικό κανόνα τη μακροοικονομία. Επίση, ε, έχουμε με νομισματική ένωση, αλλά δεν έχουμε δημοσιονομική ε, πολιτική. Οπότε, από, ε, μέσω απορρόφηση των κρατασμών γίνονται απλώ οι μισθοί, κάτι που είναι απαράδεκτο. Χρειαζόμαστε βέβαια διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά αυτές μειώνουν ακόμη περισσότερο την ιδιωτική ζήτηση. Κάτι που σημαίνει ότι είναι διασπάθηση των πόρων για αύξηση της φορολογικής εξάπλωσης μερικών χωρών, ενώ σε μερικές άλλες ε, περικόπτονται οι μισθοί και οι Μακροοικονομικά λοιπόν το αποτέλεσμα δεν θα είναι το επιθυμητό και πολιτικά θα γίνει κακή χρησιμοποίησή του. Χρειαζόμαστε πάντως δημόσιες επενδύσεις και βλέπουμε ε, σε χώρες όπως η ε, Ελλάδα που έχουν μειώσει το μισθολογικό κόστος ε, δεν έχει ξεκινήσει ανάπτυξη, γιατί η ανταγωνιστικότητα δεν αφορά μόνο την ανταγωνιστικότητα των τιμών, ε, που προέρχεται και από τους χαμηλούς μισθούς, αλλά σχετίζεται και με την παραγωγικότητα. Για την παραγωγικότητα χρειαζόμαστε επενδύσεις. Οπότε, είτε θα πρέπει να χαλαρώσουμε κάπου στους περιορισμούς στα κράτη-μέλη ίσως ε, να έχουμε ένα χρυσό κανόνα των δημόσιων επενδύσεων, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να επεκτείνουν ε, τις, ε, τις δημόσιες επενδύσεις ή να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες της ΕΤΕ ή ένα ταμείο που θα χρηματοδοτεί τέτοιες επενδύσεις. Επίσης, στην διαδικασία α, χρηματοοικονομικής των μακροοικονομικών υπηρεσιών, θα πρέπει να προσέξουμε. Μερικές πολιτικές θα πρέπει να διορθώσουν τις πολιτικές τους, ε, του υπερβολικού ελλείμματος ειδικώ, ώστε να μην χρειαζόμαστε πάρα πολλές μεταφορές. Και για να μειώσουμε τις ανισορροπίες, ε, είναι να δούμε και τι γίνεται με τις χώρες που έχουν πλεόνασμα. Κάτι που δεν έγινε στο παρελθόν. Θα πρέπει να υπάρχει στενός σύνδεσμος μεταξύ της δημοσιονομικής ικανότητας και της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Επίσης πιστεύω ότι αν θέλουμε να επιβαρύνουμε ε, υπερβολικά ένα σύστημα ε, επιδομάτων ενεργείας ευρωπαϊκού επίπεδου, χρειαζόμαστε πολιτικές που να αποκαθιστούν την πλήρη απασχόληση, κάτι που προποθέτει προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, κυρίως για να αντιμετωπιστεί η ενέργεια των νέων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Ερνέστ Μαραγκάλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος της πρώτης φάσης ε, της έκθεσης και ε, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε εν ζωή. Δεν τα έχουμε ακόμη φτύσει, κάτι που δεν είναι καθόλου αρνητικό, είναι πολύ ενθαρρυντικό. Συγχαίρω τους δύο συνεισηγητές και χαιρόμαστε για την χθεσινή και τη σημερινή ευκαιρία που έχουμε για να συμπληρώσουμε ε, το πλαίσιο και για να προσδιορίσουμε και να καθορίσουμε προτάσεις και επιλογές. Χθες οι Υπουργοί Οικονομικών το πιο σημαντικό που είπαν είναι ότι το σημείωσαν και δεν είναι πια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που το προβάλλει. Χθες ακόμη και αν ήταν λυπής η παρουσία του Συμβουλίου φάνηκε η αποδοχή της έννοιας ε, της δημοσιονομικής ικανότητας. Μπήκε πια στην ημερήσια διάταξη και στα τρία θετισμικά όργανα και αυτό είναι πολύ σημαντικό ότι άρχισαν, άρχισαν όλοι να το συζητούν. Και με τον καθηγητή Μόντι είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την ρεαλιστική και συνετή του προσέγγιση και παρουσίαση, αλλά και κάποιες νότες αισιοδοξία και ελπίδας. Οπότε ίσως τα πρώτα συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να αντιλήσουμε από ε, τις τρεις πηγές αυτές, το δικό μας έργο και τις χθεσινέ και σημερινή συνεδρίαση είναι να ολοκληρώσουμε πια τη φάση των πολιτικών πολι... Ε, των πολιτικών λιτότητας χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα για τις χώρες με χαμηλή ζήτηση. Μπορούμε επιτέλους ε, να πούμε ότι ε, ο κόσμος έχει επιδίσει, η λιτότητα δεν μας έχει οδηγήσει πουθενά και μας έχουν μείνει μόνο τα αντιπαραγωγικά και αρνητικά αποτελέσματά της με κάποια προφανή αποτελέσματα που το επιβεβαιώνουν από τη χθεσινή συνεδρίαση με τους ε, υπουργούς αλλά και στην έκθεσή μας φαίνεται η έννοια της δημόσιας επένδυσης των δημοσίων ευρωπαϊκών επενδύσεων ως βασικό στοιχείο που θα πρέπει να χαρακτηρίζει την έκθεσή μας και ε, ευρωπαϊκές δημόσιες επενδύσεις που θα πρέπει να, χρησιμο... στηρίζονται στον προϋπολογισμό αλλά και στις πιθανές συνετές εισφορές των κρατών μελών ή των νέων φορολογικών ε, δημιουργημάτων μας και ε, μια διαχείριση του χρέους που θα εξασφαλίζεται με ε, πόρους, είτε νέους είτε υφιστάμενους, που δεν θα δημιουργούν σημαντικές αλλαγές στα δημοσιονομικά επίπεδα, είτε στα εθνικά είτε στο ευρωπαϊκό. Και αυτό είναι σχεδόν κατά γράμμα, όχι αυτό που είχαμε μόνο προτείνει εμείς, αλλά και αυτό που προτείνει στην έκθεσή του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μα το είπε και η κυρία Μπέρε. Και είναι σαφώς προσδιορισμένη η κατάσταση της διεκθέσει. Το θέμα θα είναι, εμείς στη δική μας έκθεση ε, θα δώσουμε κάποιο περιθώριο σε αυτόν τον τρίτο δρόμο, πέραν του Rainy Day Fund και δηλαδή του Ταμείου Πρόβλεπτων Αναγκών και τη ανάγκη Ευρωπαϊκού Συστήματος Επιδομάτων Ενεργείας, που μα βρίσκουν σύμφωνα, Επίση και αυτά που μα είπε ο κύριο Μόντε το ήταν πολύ σημαντικά θα πρέπει να δούμε ε, σε τι θα δοθούν τα δημόσια κονδύλια αν επιμείνουμε στην ανάγκη αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Τι θα χρηματοδοτήσουν. Επίσης, το θέμα της ασφάλειας και της άμυνας είναι το πιο εμφανές παράδειγμα του ευρωπαϊκού δημοσίου αγαθού. Μας ενδιαφέρει όμως και η ενεργειακή μετάβαση, οι κλιματικές αλλαγές, η ε, κοινωνική σύγκληση, η παιδεία, η κατάρτιση, η απασχόληση σημαντικές προτεραιότητες. Έχουμε όλο το καλοκαίρι να σκεφτούμε τα θέματα και όλο το φθινόπωρο για να σκουμποθούμε, να εργαστούμε και να λάβουμε και αποφάσεις. Ευχαριστώ κύριος Εκχαουτ. ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το οποίο ελπίζω είναι όταν κάνουμε τη συζήτηση αυτή να είναι μια δεκτική συζήτηση, ανοιχτή συζήτηση και να αφήσουμε την ιδεολειψία μας την πολιτική πίσω το δεν αρκεί βέβαια να λέμε ότι αν συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις και αποκαταστήσουμε την ανταγωνιστικότητα όλο θα πάνε καλά. Δεν, τώρα ποιον κοροϊδεύεται. Νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στους λεγόμενες τρους πυλώνες. Όταν μιλάμε για τη σύγκληση στο εσωτερικό της Ευρωζώνης είναι σαφές ότι απαιτείται βέβαια να μιλήσουμε για μεταρρυθμίσεις και διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Παρ' όλα αυτά να συζητήσουμε επίσης γιατί στην παρούσα φάση οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται με συμμετρικό τρόπο. Γιατί οι πλεονασματικές χώρες δεν έχουν την ίδια στάση με τις ελληματικές χώρες. Η σύγκληση για να υπάρξει πρέπει να έρθει και από τις δύο πλευρές, γιατί αλλιώς δεν είναι σύγκληση. Όταν μιλάμε για τις ασυμματρικές συγκρούσεις, ξέρουμε ότι το πρόβλημα είναι οι επενδύσεις. Ξέρουμε επίσης ότι η πιστοτική ένωση πρέπει να ολοκληρωθεί. Αλλά μην νομίζουμε και να μην δίνουμε την εντύπωση ότι κάτι τέτοιο είναι εύκολο. Όταν μιλάμε για την Τραπεζική Ένωση, μιλάμε ας πούμε για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα εγγυήσεων, το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Ας μην κάνουμε λοιπόν σαν να είναι δεδομένη η πιστοτική αυτή ε, ένωση. Και έχουμε και τα συμμετρικά ή ασύμετρα σοκ. Όταν γνωρίζουμε ότι οι νομισματικές πολιτικές δεν έχουν καμία σχέση με αυτά και οι φορολογικές δεν παίζουν και κανένα σημαντικό ρόλο όταν ξέρουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του για τον κίνδυνο. Τότε απαιτείται να υπάρξει κάτι που δεν έχουμε και δεν έχει νόημα λοιπόν να βάζουμε προϋποθέσεις συνεχώς. Όταν συζητάμε λοιπόν ένα ταμείο για την κακιά στιγμή ή για την βροχερή μέρα όπως λέμε στα αγγλικά, ε, να μην νομίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το μέσο μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι πάντα διαθέσιμο και δεν σημαίνει ότι είναι πάντα αποτελεσματικό αυτό το Ταμείο για τις απρόβλεπτες ανάγκες. Το θέμα είναι λοιπόν πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό το Ταμείο και προσπαθούμε να διακρίνουμε διαφορετικές μορφές συνεισφοράς. Πρέπει να υπάρχει μια συνεισφορά σε αυτό το ταμείο αντικυκλική, έτσι ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιμες πιστώσεις και μέσω των τροπολογιών μας και εκτός αυτών θα πρέπει να δούμε τι κίνητρα μπορούμε να δώσουμε για τις συνεισφορές αυτές, βλέποντας ας πούμε και το θέμα της μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης των μικρό ανισοτήτων που μπορεί να υπάρχουν. Προσπαθήσαμε επίσης ε, στις προτάσεις μας να βάλουμε και μία κατά κάποιο τρόπο ρήτρα προστασίας. Αν δούμε ότι κάποιες χώρες οποφελούνται επί υπερβολικά, η τροπολογία 661. Υπάρχει και ο λεγόμενος δεοντολογικός κίνδυνος Εν πάση περιπτώσει ας σταματήσουμε όμως να εμένουμε στη μοναδικότητα των μεταρρυθμίσεων. Είναι κουραστικό. Νομίζω ότι πάντα έχει σημασία να υπάρχει επίσης και ένα ανώτατο όριο σε σχέση με τις δημοσιονομικές ικανότητες. Η αιρεσιμότητα από μόνη της δεν αρχεί, α, χρειάζεται ακριβώς αυτό το όριο. Τότε μόνο θα έχουμε σύγκληση, τότε θα έχουμε την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τα συμμετρικά σοκ, πόσο μάλλον δεν τα ασύμετρα. Ας ξεπεράσουμε τις ιδεολειψίες μας και ας κάνουμε μια ευφυή συζήτηση, να κάνουμε ευφυείς προτάσεις και αυτό να γίνει και σε εθνικό επίπεδο. Εγώ δεν θα έλεγα, έχω πολλές πολλή εμπιστοσύνη για αυτές τις μεγάλες συναντήσεις που κάνουμε στις Βρυξέλλες. Οι συζητήσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν στα εθνικά κοινοβούλια, γιατί αλλιώς θα παραμείνουν σε θεωρητικό επίπεδο και δεν πρέπει. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σωστά, Μάρκο Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές όπως ακριβώς φάνηκε και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ανάμεσα στους σκιώδεις, εγώ δεν συμμερίζομαι την πρόταση αυτή και δεν συμμερίζομαι την εμπιστοσύνη που έχουμε στο μέσο αυτό σαν κάτι το οποίο θα αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού για τα προβλήματα της Ευρωζώνης. Ιδιαίτερα με τη μορφή που παίρνει και το σχέδιο να υπάρξει μια δημοσιονομική, αν θέλετε, αυτονομία για την Ευρωζώνη. Δεν μ' αρέσει αυτό. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ένα τέτοιο μέσο δεν πρόκειται να επιλύσει τις μακροοικονομικές ανισότητες που προκλήθηκαν από, την, από το ενιαίο νόμισμα στην Ευρωζώνη. δεν μπορούμε να αγνοήσουμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια α, θεωρίας οικονομικής για τις νομισματικές περιοχές, ενωμένες νομισματικά περιοχές κτλ. Σαν την Ευρωζώνη. Βλέπουμε στην έκθεση ότι πάρα πολύ συχνά γίνεται αναφορά για ένα σύστημα μεταφορών που δεν θα πρέπει να είναι μόνιμο, και αν η Ευρωζώνη θέλει να λειτουργήσει καλύτερα από σήμερα, αυτό το οποίο έχει ανάγκη είναι οι μόνιμες μεταφορές, οι οποίες απ' την άλλη πολιτικά είναι προβληματικές. Έχουμε σήμερα δύο μεγάλες χώρες της Ευρωζώνης με εκλογές το 2017 και είναι πάρα πολύ δύσκολο, εγώ φαντάζομαι τη Μέρκελ να κάνει προεκλογική εκστρατεία, λέγοντας ότι για να γίνει πιο βιώσιμη η Ευρωζώνη η Γερμανία θα πρέπει να μεταφέρει 150 ή 200 δις ευρώ σε αιτήσια βάση προς την περιφέρεια. Οι Γερμανοί φίλοι το γνωρίζουν όμως ότι αυτό το οποίο σημαίνει συνέβη όταν επανενώθηκε η Γερμανία ακόμα και τώρα τα πέντε λέντερ της Ανατολικής Γερμανίας ε, ζουν κάτω από, μόνιμες, ε, από καθεστώς μόνιμης μεταφοράς ρευστότητας από τη Δύση. Δεν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ένα μέσο το οποίο θα καταστήσει αμέσως λειτουργική την Ευρωζώνη. Κάποια άλλα ανησυχητικά σημεία τα οποία βλέπω είναι η λεγόμενη θεσμικοποίηση ακριβώς του μηχανισμού παρέμβασης και σταθεροποίησης των οικονομιών. Το να θελήσει κανείς να μετατρέψει τον μηχανισμό αυτό σε ένα μόνιμο ευρωπαϊκό ταμείο είναι κάτι το οποίο βρίσκω εγώ σαν επικίνδυνο και νομίζω ότι έχει άμεση σχέση και με την απαράδεκτη και αποτυχημένη διαχείριση από πλευράς της Τρόικα προβλημάτων όπως το ελληνικό και οι πολιτικές του Δέλτα Νιτάφ επίσης, οι οποίες και στο εσωτερικό της Ευρωζώνης όπως και σε άλλες χώρες εκτός Ένωσης απέτυχε και γι' αυτό ακριβώς τέτοιου είδους λογικές και για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δέλτα Νιτάφ δεν με ικανοποιούν και με ανησυχούν. Αυτό το οποίο έχει ανάγκη πραγματικά η Ευρωζώνη είναι κάτι το πάρα πολύ απλό και εδώ θα ήθελα στην προσπάθεια της αναζήτησής μας να το συζητήσουμε. Θα πρέπει να αφήσουμε επίσης ε, να υπάρξουν διακυμάνσεις ε, στις ε, συναλλαγματικές ισοτιμίες ανάμεσα στις διαφορετικές χώρες εκτός Ευρωζώνης και να δούμε τι θα κάνουμε και με τους κανόνες του Μάστριχτ που έχει παράλογους ε, κανόνες που καταστρέφουν την πραγματική Ευρώπη. Αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα στην Ευρώπη είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων στην έρευνα, στην εκπαίδευση κτλ. Οι κανόνες λοιπόν του Μάστριχτ είναι παράλογοι και μπλοκάρουν τις χώρες και δεν τους επιτρέπουν να προχωρήσουν ε, στην πρόοδο. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την ομάδα ΕΝΕΦ. Είναι κανείς εδώ? Όχι. Ωραία, περνάμε στο Catch the Eye. Ο κύριος Χόκμαρ είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι το σωστό σημείο εστίασης είναι πώς να αποφύγουμε τα διάφορα είδη κρίσεων και αυτό βέβαια υπογραμμίζει ε, την ανάγκη εντοπισμού του βασικού προβλήματος που είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Όχι η έλλειψη ε, κονδυλίων που καλύπτουν τα σφάλματα που έχουν κάνει οι κυβερνήσεις ε, μη αναδιαρθρώνοντας τις οικονομίες τους. Και πρέπει να πω ότι αν δούμε, κανείς, αν τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής ευρωπαϊκής οικονομίας έχουμε 10 με 15% ε, φορολογικό βάρος από οποιαδήποτε άλλη ανταγωνιστική περιφέρεια. Και αυτό πλήττει το επενδυτικό κλίμα. Το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά. Ξέρουμε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις χάνουν έδαφος, ξέρουμε ότι το επιχειρηματικό κεφάλαιο χάνει έδαφος και πρέπει αυτό να αντιμετωπίσουμε, όχι να αυξήσουμε τους, δημο... τους... Ε, το... τον προϋπολογισμό ε, για τις δημόσιες δαπάνες. Αυτό ε, είναι κάτι που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Υπάρχει μια ισχυρή δημοσιονομική ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά, αυτή είναι οι προϋπολογισμοί των κρατών μελών. Και το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις που έχουν ε, ε, λάθος ερμηνεύσει το σύμφωνο σταθερότητας και νομίζουν ότι ε, το μείον 3 είναι ε, το, κατώτατο, το ανώτατο όριο. Όχι, είναι το κατώτατο και πρέπει να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε αυτή την ικανότητα για να αντιμετωπίσουμε τις δύσκολες ώρες. Και αυτή η ικανότητα είναι πολύ μεγαλύτερη αν προγραμματίζεται με το σωστό τρόπο και δεν νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι μπορούμε να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με νέους θεσμούς και νέους κανόνες νομίζω ότι πρέπει να βασιστούμε στους υφιστάμενους κανόνες και θεσμούς έχουμε μια δημοσιονομική ικανότητα και ονομάζεται ε, σύμφωνο σταθερότητας Ευχαριστώ Η Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Χθες ο Σλοβάκος ε, Υπουργός Καζίμιρ είπε ότι όταν μιλούμε για δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει πρώτα να προσδιορίσουμε τα μέσα και μετά να δούμε πώς θα τα χρηματοδοτήσουμε. Εν μέρη συμφωνώ μαζί του. Και όντως θα πρέπει να τα καθορίσουμε όλα αυτά με σαφήνεια για να δούμε τι είδους χρηματοδότηση θέλουμε για τα μέσα που έχουμε συμφωνήσει. Αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ στη συζήτηση αν δεν, έχουμε, αν δεν σκεφτόμαστε σχεδόν παράλληλα και τη χρηματοδότηση. Γιατί θα έχουμε απλώς ιδέες και ίσως ουτοπίες, ε, αλλά δεν θα μπορούμε να τις χρηματοδοτήσουμε αν δεν έχουμε ε, κονδύλια, ή πηγές χρηματοδότησης. Στην έκθεση Μπέγκε Μπερές θα, θα πρέπει τουλάχιστον από πλευράς προπολογισμού να προτείνουμε κάποια χαρακτηριστικά ή κάποιες βασικές ε, γραμμές ε, κατευθυντήρες που θα πρέπει να ακολουθεί, από αυτές θα πρέπει να διέπεται η δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης. Και αν θέλουμε ο προπολογισμό τη Ευρωζώνη να συμπεριλαμβάνεται στο γενικό προπολογισμό τη Ένωση θα πρέπει να είναι εκτό του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου. Αυτό είναι βασική κατευθυντήρια γραμμή. Δεύτερον, θα πρέπει να χρηματοδοτείται με ίδιου πόρου. Αλλιώ θα ε, προσκρούσουμε στο ανώτατο όριο των δαπανών του 1,29 και θα πρέπει όλα αυτά τα χρηματοδοτήσουμε το 0,3 του ΑΕΠ. Και επίσης θα πρέπει να πρόκειται για νέο χρήμα, φρέσκο χρήμα, δηλαδή για να μην ενδίδουμε στον πειρασμό να ε, προσπαθούμε να παίρνουμε από μερικά τμήματα του προπολογισμού της Ένωσης και να να χρηματοδοτούμε κάποιες πολιτικές ευρωζώνης. Αυτά από δημοσιονομική άποψη. Τώρα πιο γενικά υπό τη σκοπιά της ΕΚΟΝ. Ε, κάποιος μας μίλησε για μάντρα, για εποδούς, εγώ θα μιλήσω για μύθους. Και παρόλο που προσπαθούμε να τους καταρρύψουμε αυτούς τους μύθους, εξακολουθούν να ισχύουν. Ε, οι κανόνες, αν ε, τηρηθούν οι κανόνες, αν τηρηθούν τα κριτήρια του Μάστριχτ, ε, είστε στο πυρόβλητο. Όχι, δεν ισχύει αυτό και είμαστε η Ισπανία χαρακτηριστικό παράδειγμα, που είμαστε οι καλύτεροι μαθητές ε, των κριτήριων του Μάστριχτ. Χρέος κάτω του 60% δεν είναι ότι είχαμε έλλειμμα, είχαμε ε, πλεόνασμα. Και λίγα χρόνια μετά βλέπετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Επίση, διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Ανατριχιάζω κάθε φορά που ακούω αυτή τη λέξη, γιατί μα παρουσιάζονται ω η πανάκια όλων των προβλημάτων και κανένα δεν ε, δίνει το σωστό χαρακτηριστικό σε αυτέ τι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Μπορεί να είναι καλέ και κακέ ανάλογα με του ε, αλλά ε, τι είδου διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει. Νομίζω ότι μα περισσεύουν οι διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσει παρά μα λείπουν. Αλλά γιατί στόχου και τι είδου μεταρρυθμίσει θέλουμε. Και επίση ε, οι συνταγέ που εφαρμόζουμε. Από το 2008 που ξέσπασε η κρίση έχουν περάσει 8 ε, χρόνια και τα μέτρα που έχουμε εφαρμόσει δεν έχουν αποδώσει. Κάποια χαμηλή ανάπτυξη αλλά με αύξηση ε, του χρέους, ε, μεγαλύτερες ανισορροπίες και ανισότητες από το 2008. Θα πρέπει λοιπόν να αντιστρέψουμε όλες τις πολιτικές της τελευταίας οκταετίας. Και αυτό δεν είναι ποδός, δεν είναι ούτε μύθος, απλώς είναι ενυφάλια διαπίστωση των αποτελεσμάτων των πολιτικών μας της τελευταίας οκταετίας. Ευχαριστώ. Μάριος Ροζάτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχουν τρει λόγοι που αναφέρονται στην έκθεση σε ό,τι αφορά τη δημοσιονομική ικανότητα στην Ευρωζώνη. Το πρώτο, ο πρώτο λόγο είναι τα ασύμετρα σοκ. Αν υπάρχει ένα κρατό μέλο στην Ευρωζώνη το οποίο χτυπήθηκε από ένα τέτοιο ασύμετρο σοκ, η ιδέα και η, η όλη ιδέα της δημιουργία τη Ευρωζώνη ήταν ότι θα μπορούσε η χώρα αυτή να αντιδράσει με δημοσιονομική πολιτική, όχι με νομισματική πολιτική ασφαλώ. Κοιτώντα όμω αυτά τα σύμμετρα σοκ και συμφωνώ με όσου ανέφεραν ότι δεν ήταν τόσο ασύμμετρα τελικά αυτά τα σοκ και να μην τα συγχαίω με αυτά με έλλειψη σύγκληση γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Αλλά κοιτώντα τα ασύμμετρα σοκ στην Ευρωζώνη βλέπουμε ότι χτύπησε κυρίω χώρε που δεν είχαν δημοσιονομικό περιθώριο εξ αρχή είχαν δηλαδή ελλείμματα πολύ κάτω του 3% και δεν μπορούσαν να μειώσουν τις δαπάνες τους και παράλληλα είχαν και υψηλό χρέο. Άρα ε, στην περίπτωση αυτή ασφαλώς και αναζητήσαν άλλα μέσα, ίσως και τη δημοσιονομική ικανότητα. Αλλά ο λόγος της κρίσης, ε, η αιτία της κρίσης ήταν στις χώρες αυτές η έλλειψη αυτού του δημοσιονομικού περιθωρίου και αυτό επειδή δεν είχαν τηρήσει τους κανόνες για το χρέος και το έλλειμμα. Αν δεν ε, λοιπόν λύσουμε το θέμα αυτό και περάσουμε κατευθείαν στη δημοσιονομική ικανότητα, τι θα γίνει, θα ξεχάσουμε τα αίτια, τα βαθύτερα αίτια της κρίσης και ακόμα κι αν ε, δημιουργηθεί η δημοσιονομική ικανότητα. Θα βρεθούμε στην κατάσταση όπου οι χώρε αυτέ οι οποίε παραβίαζαν του κανόνε στο παρελθόν θα συνεχίσουν τον πράγμα αυτό στο μέλλον. Και τι νόημα έχει τότε να υπάρχει μια δημοσιονομική τέτοια ικανότητα η οποία θα καταλήξει σε μια ε, μονοδρομή μεταφορά πόρων προς τις χώρες αυτές που δεν τηρούν τους κανόνους. Αυτό για τα σύμμετρα σοκ. Τώρα το δεύτερο, μίλησατε για τα κίνητρα για τις διευθυντικές μεταρρυθμίσεις. Και εδώ θεωρώ ότι είναι μεγάλος ο κίνδυνος του ηθικού ρίσκου. Τι νόημα έχει να δίνονται κίνητρα για τα κράτη-μέλη για να κάνουν διευθυντικές μεταρρυθμίσεις προς όφελος του κράτους μέλους. Το ίδιο ουσιαστικά τα κράτη-μέλη θα περιμένουν. Θα περιμένουν μέχρι να πάρουν κάποια χρήματα τα οποία θα τους ε, χρησιμεύσουν για το καλό της χώρας. Πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν αυτό τον ηθικό κίνδυνο, αυτό τον κίνητρο διόνυσης των προβλημάτων. Ένα τρίτο θέμα, το θέμα της εγγύησης για την ανεργία. Αν υπάρχει υπερβολική ανεργία σε κάποιο κράτος μέλος, αυτό προκαλείται από δύο λόγους, είτε κυκλικούς λόγους, ύφεση, αλλά στην περίπτωση αυτή πάλι επανερχόμαστε στο θέμα της δημοσιονομικής πολιτικής. Θα πρέπει να υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο για να δοθούν απαντήσεις. Αν δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο γιατί υπάρχει υπερχρέωση, ασφαλώς η χώρα αντιμετωπίζει προβλήματα. Η επίλυση όμως του προβλήματος δεν είναι η δημοσιονομική ικανότητα, αλλά η τακτοποίηση των δημοσιονομικών λογαριασμών. Και υπάρχει και ένα δεύτερο λόγο που προκαλεί ανεργία. Διαρθωτική λόγοι. Πολύ απλά είναι τόσο άκαμπτη η αγορά εργασία που τελικά η χώρα πλήττεται διαρκώ από ανεργία. Και πάλι όμω η λύση είναι οι διαθωτικές μεταρρυθμίσει στην αγορά εργασία, προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη. Καταλαβαίνω ότι αυτό ενδεχομένω για κάποιου είναι ανέφικτο, αλλά αυτό είναι το μάντρα το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε στο σημείο αυτό. Δεν είμαι αντίθετος με όσους είναι για το, τη δημοσιονομική ικανότητα. Δεν είμαι επί τη αρχής κατά. Αλλά πιστεύω ότι αποτελεί επιταγή να κοιτάξουμε καταρχάς γιατί δεν τηρήθηκαν οι δημοσιονομικοί κανόνε και να διορθώσουμε κατά δεύτερον την κατάσταση αυτή. Όπου τα κράτη-μέλη δεν μπορούν ή δεν θέλουν να τηρήσουν του δημοσιονομικού κανόνε Και μόνο αν δούμε στη συνέχεια ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες γιατί οι χώρες παρά το γεγονός ότι έχουν περιθώρια 3-4% στους προϋπολογισμούς τους πλέον χρειάζονται ακόμα κίνητρα για την οικονομία τους και ακόμα υπόκεινται ασύμετρα σοκ. Εκεί να κοιτάξουμε την δημοσιονομική ικανότητα, αλλά παράλληλα με άλλα μέσα, όπως είναι για παράδειγμα ο μηχανισμός ιδιωτικής κατανομής του κινδύνου. Δεν συζητήθηκε μια πλήρης τραπεζική ένωση ή κεφαλαϊκή ένωση. Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή, ο οποίος και μίλησε πέντε λεπτά. Ο κ. Λεβαντόφσκι έχει το λόγο. Δεν θέλω να επαναλάβω, γιατί είναι σημαντική η συλλογική ευθεία. Υπάρχει μία κρυμμένη υπόθεση πριν από, πίσω από την ιδέα της δημοσιονομικής ικανότητας της Ευρωζώνης ε, και αυτή η υπόθεση είναι ότι δεν είναι δυνατόν ε, να ε, επιβάλλουμε την συμμόρφωση με τους συμπεφωνημένους κανόνες, τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωζώνης και επίσης ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν αρκετή γενναιότητα ώστε να αναλάβουν το πολιτικό ε, κόστος ε, για τις ε, πολύ δύσκολες και δαπανηρές αλλαγές στο, στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι κάτι ε, που εμένα δεν με έχει κουράσει. Δεν με έχει κουράσει η εποδός των διαρθρωτικών αλλαγών αν είναι αμφίδρομη, ε, είτε είναι κακή η επίδοση, που αυτό είναι ένα σημείο ε, αναφοράς, ή αν υπάρχει κάποιο είδους συγκριτική αξιολόγηση άλλων ε, χωρών, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, ε, που δεν είναι έτοιμες ε, να αναλάβουν το πολιτικό κόστος διαρθρωτικών αλλαγών. Αν αυτή είναι η υπόθεση πίσω από τη δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης, αυτό σημαίνει ότι ο ηθικός κίνδυνος είναι αναπόφευκτος. Θα βρεθούμε ενώπιον αυτής της κατάστασης, γιατί δημιουργούμε ένα δημοσιονομικό κίνητρο ε, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μεταρρυθμίσεις που είναι πολύ σημαντικές στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Πριν δώσω το λόγο ε, στους εισηγητές, ε, θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Χόκμαρκ, ο οποίος όμως αποχώρησε. Παρ' όλα αυτά θα του απαντήσω. Είναι μεγάλη η διαφορά του να είναι κανείς στην νομισματική ένωση ε, ή να μην είναι, γιατί όταν είναι κανείς ε, ε, γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει σε σχέση με τη συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι το οποίο δεν ισχύει στην άλλη περίπτωση. Αυτό το οποίο αναφέρεται στην έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το χαρακτηριστικό ε, που αρχικά είχε εντοπιστεί αυτής ε, ε, για αυτήν την δημοσιονομική ικανότητα είναι ότι θα έχουμε μια νομισματική πολιτική η οποία θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ε, τα συμμετρικά σοκ και την εθνική πολιτική, τη δημοσιονομική πολιτική για τα συμμετρικά σοκ. Όμως το πολιτικό επιχείρημα είναι ότι από τη μία υπάρχει πολύ έντονη κριτική ότι φτάνουμε στα όρια μας ή ενδεχομένως πήγαμε και πολύ μακριά με το πώς αντιμετωπίσαμε τις κρίσεις, ε, κάτι το οποίο δεν ήταν αυτό που είχαμε αρχικά ε, ε, σκεφτεί όταν είδαμε για παράδειγμα πώς η νομισματική πολιτική μπορεί να αντιμετωπίσει ένα συμμετρικό σοκ, μια συμμετρική κρίση. Μπορούμε να πάμε πολύ ε, πέρα από αυτό το οποίο θέτουν ένα αμφιβόλο ε, ορισμένοι. Επίσης υπάρχει και ο περιορισμός της δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους. Πάντως είναι σαφές ότι πρέπει να έχουμε ε, συγκεκριμένους, ε, συγκεκριμένους περιορισμούς ε, για τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την αντιμετώπιση των ασυμμετρικών κρίσεων. Είναι λοιπόν δύσκολο να πει κανείς, να ισχυριστεί κανείς ότι δεν έχουμε ένα ιδανικό μοντέλο και ότι έχουμε ήδη κάποια ε, εργαλεία στη διάθεσή μας. Έχουμε ε, μία ισχυρή δημοσιονομική ε, πολιτική, εκτός αν λέτε ότι δεν χρειαζόμαστε καθόλου το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, εκτός αν θέλετε ένα τελείως διαφορετικό εργαλείο όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να αμφισβητήσει κανείς τη βασική ε, ιδέα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολιτικές δυσκολίες, οι δυσκολίες της μετάβασης, σε τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία νομίζω ότι αναφέρονται στην έκθεση και πολλές τροπολογίες το καλύπτουν, ε, πώς μπορεί ε, κανείς να έχει μία προσέγγιση, να βασιστεί κανείς στον υπάρχοντα προϋπολογισμό, να αρχίσει με μία περιορισμένη δημοσιονομική ικανότητα, και σιγά σιγά να την ξεπεράσει. Ε, αναφέρθηκε ήδη αυτό, δεν χρειάζεται να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, όμως... Ε, αυτό ε, που ζητήσατε να μην υπάρξει ιδεολογική συζήτηση ε, για τα βασικά, για τα στοιχειώδη, ε, δεν βρήκε σύμφωνους άλλους, άλλους ομιλητές, όμως εγώ θα ήθελα να ενθαρρύνω τους εισηγητές να έχουν μια ρεαλιστική και επικοδομητική προσέγγιση, γιατί αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση για να αντιμετωπίσουμε βασική ιδεολογία της οικονομικής πολιτικής, δεν ε, ε, θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη ε, η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και σας συνιστώ να τη διαβάσετε προσεκτικά. Να δώσω τώρα τον λόγο στους εισηγητές. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο πρώτος. Περβόνς. Ευχαριστώ πολύ. Δεν, είμαστε, δεν έχουμε μείνει και πάρα πολύ. Έχει περάσει η ώρα και θα είμαι πολύ σύντομη. Πριν μπω στις λεπτομέρειες της απάντησης, θα ήθελα να πω κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση. Κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει ότι βιώνουμε μία περίοδο έντασης και αμφιβολίας στην Ευρώπη. Κάτω από τέτοιου είδους συνθήκες η Ευρώπη έχει σημειώσει στο παρελθόν βήματα πρόοδου. Η... Την Τραπεζική Ένωση κάναμε αυτό το άλμα γιατί βιώναμε μία κρίση και αυτή η κρίση όταν βλέπουμε το επίπεδο επενδύσεων στις οικονομίες μας, την έλλειψη σύγκλησης και το σοκ το οποίο προκαλείται σε ό,τι κάνουμε το αποτέλεσμα του Βρετανικού δημοψηφίσματος μας οδηγεί στη διαπίστωση ότι ζούμε μία κρίση. Λοιπόν, δεν είναι σωστή η αντίδρασή του, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα για να μην σπάσουμε και άλλα αυγά. Αντίθετα, πρέπει να κάνουμε ένα ακόμη βήμα και να αναλάβουμε την ευθύνη μας για την επόμενη φάση, κάτι το οποίο αρνούμεθα να κάνουμε εδώ και πολύ καιρό και αυτό το περιλαμβάνεται και στο πακέτο του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ. Τώρα σε σχέση με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μουρεσάν για το moral hazard. Τι νόημα έχει μια χώρα όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα να μην κάνουν μεταρρυθμίσεις για να βρεθούν στο τέλος κάτω από εντολή της Τρόικα με μια ιδιαιτέρως περιορισμένη κυριαρχία και με ελάχιστα περιθώρια κίνησης. Δεν υπάρχει αυτή η λύση. Δεν είναι λοιπόν λόγο moral hazard, δεν είναι λόγο μη σεβασμού των κανόνων. Δεν έγιναν σεβαστοί οι κανόνες γιατί δεν ήταν προσαρμοσμένοι και δεν έλαβαν υπόψη τους την πολλαπλότητα των οικονομιών της Ευρώπης, όπως και την δυναμική που δημιούργησε το ίδιο το ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν πράγματι θέλουμε να ξεπεράσουμε τη λύση αυτή, την κατάσταση αυτή, την οποία και εγώ συχαίνομαι, γιατί και εγώ πιστεύω ότι οι οικονομίες μας πρέπει να μεταρρυθμιστούν. Αλλά από ό,τι φαίνεται με το σύμφωνο σταθερότητας δεν έχουμε βρει ακόμα τον σωστό οδηγό. Και καταλαβαίνω να τίθεται το θέμα του moral hazard βέβαια. Όπως μας είπε και ο Μπενουά Κερέ, όταν είχαμε οργανώσει την προηγούμενη ακρόαση, λόγω του κινδύνου του moral hazard, στην ουσία απαγορεύουμε κάθε μορφή πρόοδου. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό και διευρύνουμε και τον κίνδυνο αυτό για να απαγορεύσουμε κάθε εξέλιξη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση οδηγούμεθα στην καταστροφή. Δεν κάνουμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα να γίνουν. Ε, αυτά που είπε τώρα ο Ντάριος Ροζάτη για το αν είναι συμμετρικά ή μη τα σοκ. Νομίζω ότι έχω ήδη απαντήσει σε αυτό, ε, Ντάριος, όταν συζητήσαμε το θέμα του βασμού των δημοσιονομικών κανόνων. Ε, πράγματι μια συμμετρική κρίση επηρεάζει τα κράτη-μέλη με ασύμετο τρόπο ανάλογα με το επίπεδο και την κατάσταση της οικονομίας της την ώρα και την οποία επισυμβαίνει. Συνεπώς λοιπόν ε, είναι κάτι αυτό που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε όταν αξιολογούμε τις οικονομίες. Όταν εμείς μιλάμε για λύσεις τις οποίες θα πρέπει να θέσουμε σε λειτουργία για να αντιμετωπίσουμε τις ασύμετρες αυτές μορφές σοκ, έχουν γίνει μέχρι τώρα δύο προτάσεις, οι οποίες υποστηρίζονται και από τους δύο ε, εισηγητές, τα λεγόμενα Rainy Day Fund, το λεγόμενο Rainy Day Fund ε, για περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης. Γιατί δεν έχει υπάρξει κάτι τέτοιο. Δεν οφείλεται αυτό στην κακή θέληση των ε, κρατών μελών, αλλά γιατί δεν μπορέσαμε να βρούμε τον δυναμισμό που θα μας επέτρεπε να θέσουμε σε λειτουργία αυτόν τον κανόνα της καλής διαχείρισης για, την, ε, για το ελάχιστο κοινό επίπεδο, επίδομα μάλλον ανεργίας. Το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε εμείς στους μηχανισμούς οι οποίοι ισχύουν στις διάφορες χώρες, αλλά θα πρέπει εμείς να αντιμετωπίσουμε ένα ασύμετρο σοκ και όταν υπάρχει μια συγκυριακή μορφή ανεργίας και όχι διαρθρωτική, και το είπε πολύ σωστά ο Τσακαλώτος χθε το απόγευμα, πως ε, μια κυκλική μορφή ανεργίας, αν δεν αντιμετωπιστεί σύντομα, μετασχηματίζεται σε διαρθρωτική ανεργία και καθίσταται σημείο επιβάρυνσης των αρνητικών προβλέψεων της οικονομίας. Λοιπόν, ε, η κυκλική ανεργία ε, θα έπρεπε να οδηγεί σε μία ελάχιστη ίσως μορφή επιδόματος Αναφέρομαι για το συγκυριακό βέβαια φαινόμενο της ανεργίας. Αν δεν το κάνουμε αυτό τότε θα επιβαρύνουμε τον φαύλο κύκλο της ευρωπαϊκής οικονομίας και όχι μόνο της χώρας η οποία κατά περίπτωση φύγεται περισσότερο. Λοιπόν, μία επιπλέον παρατήρηση ε, συμπληρώνοντας αυτά που είπε ο Φάμπιο Ντεμάζη. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι το μέσο των μακροοικονομικών ισορροπιών δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει επαρκώς και να πω στον συνάδελφο Μαραγκάη ότι και εγώ αγαπώ την ιδέα του κοινού ευρωπαϊκού αγαθού αλλά έχω ένα μικρό ερώτημα όταν βλέπω τα παραδείγματα τα οποία χρησιμοποιήσατε στον τομέα της ασφάλειας, της άμυνας, ε, και της ταύτισής της με τη ζώνη ευρώ. Εκεί ίσως να υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία πρέπει ακόμα να μας απασχολήσουν. Πάντως συμφωνώ ότι η έννοια της διακυβέρνησης ε, είναι κάτι που μπορεί να συνδεθεί με την έννοια του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος και του κοινού ευρωπαϊκού αγαθού μακρηγορώ, αλλά νομίζω ότι αυτά που λέμε ίσως να είναι χρήσιμα για την επεξεργασία συμβιβαστικών προτάσεων. Σας ευχαριστώ. Και τέλος ο κύριος Μπέγκε, για να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από την αρχή δεν το έθεσα το θέμα αυτό και δεν έκρυψα ότι θα μπορούσα να φανταστώ εξ αρχής ότι στο τέλος θα καταφέρουμε, ελπίζω, να συνεργαστούμε ε, για να συμφωνήσουμε όλοι και να αλλάξουμε τον τίτλο της έκθεσης αυτής, να μιλάμε για την σταθεροποίηση της Ευρωζώνης και τις δημοσιονομικές προκλήσεις που συνδέονται με το θέμα αυτό. Και συμφωνώ με τον συνάδελφο Ροζανάτη και Λεβαντόφσκι. Θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα όταν μιλάμε για θέματα εμπιστοσύνης, όταν αφενός έχουμε τα αναμφίβολα επιτεύγματα και τις επιτυχίες μας μέσα στην κρίση, το οποίο μας οδήγησαν και σε πολλές βελτιώσεις ε, ε, σημαντικές ε, του συστήματος. Δεν θα πρέπει αυτά να τα αγνοούμε. Και για να πω και προς, προς ένα συνάδελφο Ιταλό πιο νέο, όταν μιλάει για την δεκαετία του 70 για την Ιταλία, νομίζω ότι δεν ξέρει για το τι μιλάει. η αγορά ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης και αυτό για όλους και γι' αυτό λοιπόν ξεκίνησε η απόπειρα για το κοινό νόμισμα. Αλλά αυτά είναι ιστορίε τι οποίε δεν τι αναλαμβάνεται ο καθένα με τον ίδιο τρόπο ενδεχομένω. Και στι συζητήσει λοιπόν αυτέ, ο σκοπό ήταν να γίνει και ανάλυση για κάποια μέσα, γιατί δεν υπάρχουν ενδεχομένως προβλήματα και που είναι πολύ περίπλοκο το νομοθέτημα, τα νομοθετήματα και πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε τα πράγματα αυτά προς όφελος όλων των συμμετεχόντων. Και φυσικά, όταν στην τελική ανάλυση μιλάμε για δημοσιονομικές ικανότητες, είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει ένας παράλληλος προϋπολογισμός, δεν υπονομεύουμε τα υφιστάμενα εργαλεία για αυτά που κάνουν οι φυτικά ταμεία. Αυτό θα πρέπει να διευκρινίζεται. Και όταν μιλάμε για τον ηθικό κίνδυνο, φυσικά θα πρέπει να αποφευχθεί. Αλλιώς δεν είμαστε αξιόπιστες, αλλά δεν είμαστε και ειλικρινείς. Τα υφιστάμενα μέσα τα δημιουργήσαμε ουσιαστικά μόνο για να ξεπερνάμε και να υπερβαίνουμε τις εθνικές δραστηριότητες. Μπορούμε επίσης να συζητήσουμε κατά πόσον όλα τα project τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΦΣΥ θα είχαν έτσι κι αλλιώς πραγματοποιηθεί ε, εν μέρη, αλλά ενδεχομένω να έχει πάρει πιο πολύ χρόνο. Όλα αυτά είναι στα πλαίσια της ειλικρίνειας ε, μεταξύ μας και όχι μόνο το να συζητάμε θέματα τα δημοσιονομικής ικανότητας και ηθικού κινδύνου. Θα ήθελα λοιπόν και δεδομένη στις εμπειρίες μου να πω το εξή. Ναι, να συνεχίσουμε τις ρευτικές μεταρρυθμίσεις, μάλιστα. Ε, μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, σε κάποιες χώρες γίνεται αυτό, σε κάποιες χώρες δεν έχει γίνει αυτό επαρκώς, ε, εννοείται, αλλά παράλληλα να προσπαθήσουμε πάντα να τηρούμε ισορροπίες. Για παράδειγμα, ε, κοιτώντας τι γίνεται στη δική μου τη χώρα, σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλους τους τομείς, αλλά σε κάποιους ε, τομείς έχουμε μια καταγερματισμό της αγοράς εργασίας και δημιουργούνται θέσεις εργασίας, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες ε, νέοι, όχι μόνο ταχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, αλλά και μακροπρόθεσμα, αν δεν είμαστε στον τρόπο είναι νομοθεσία, έχουν πρόβλημα και αν δεν υπάρχει και η ισορροπία μεταξύ επιχειρησίων και συνδικάτων τελικά θα καταλήξουν να παραμείνουν ε, στα πλαίσια της επισφαλούς θέσης, στα πλαίσια της επισφαλής απασχόλησης. Έχουν θέσεις απασχόλησης, αλλά ε, μήπως ε, έχουν χρήματα, μήπως ε, ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό απλά αναβάλουμε την επίλυση του προβλήματος και μεταφέρουμε το πρόβλημα στη συλλεξιβότητα του μέλλοντος και να μην τα αλλάζουμε όλα βάθρων. Να μην ξεχνάμε επίσης και το εξή. Όταν κοιτούντας ε, τις δεσμεύσεις ε, για το φετινό έτος, αν ζητάμε από την Ελλάδα, και τα επαναλαμβάνω αυτά, αλλά θα πρέπει να τα πω και σε αυτούς τους κόλπους, όταν λέμε στην Ελλάδα ότι σε πέντε χρόνια θα πρέπει το υγρό να έχει αναμορφωθεί, να έχει αναδερθωθεί πλήρως. Και στο δικό μου όμως που το κρατήριο δεν μπορούμε να βάλουμε ένα κανάλι να φτιάξουμε για την εσωτερική αγορά. Δεν καταφέρουμε δηλαδή να φτιάξουμε αυτό το κανάλι, αυτή τη γέφυρα με τη Δανία μέσα σε 10 χρόνια. Και υπάρχουν αναβολέ, καθυστερήσει επενδύσει. Ε, μα θα πρέπει να κοιτάξουμε όλα αυτά. Γιατί υπάρχει τόσο λίγη εμπιστοσύνη και πού είναι οι κανόνε μα για τη συμμετοχή των κρατών σε επίπεδο ομόσπονδο, ομοσπονδιακό, εθνικό, ευρωπαϊκό, με την ε, επιμέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί όλα αυτά έχουν καταστεί τόσο περίπλοκα που δεν μπορούμε να τα κατανοήσει κανένα. Έχει νόημα να διαβάζουν τα βιβλία αυτά. Όλοι μας λοιπόν, όλοι μας λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε λίγο αυτοκριτική και να μην μιλάμε για μεταρρυθμίσεις τους οποίες απαιτούμε από τους πολίτες μας, κάποιες φορές είναι επώδυνες, αλλά τελικά δεν κάνουμε επαρκείς μεταρρυθμίσεις στο κράτος διευθυντικά. Και αυτό αφορά και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να μην το ξεχνάμε αυτό, αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι. Σε ό,τι αφορά το θέμα της χρηματοδότησης, νομίζω ότι υποστηρίζω αυτά που είπαν και οι συναδελφοί. Προηγουμένω, το πώ θα, θα βάλουμε πέρα στον προπολογισμό πλέον, όπου κανεί δεν ξέρει τι θα σημαίνει το Brexit για την αναθεώρηση αν θα είναι παράλληλη αυτή η διαδικασία, αν θα αναβληθεί, βρισκόμαστε πραγματικά σε μια φάση περιπέτειας και θα πρέπει ρεαλιστικά να κοιτάξουμε τα μέτρα με τα οποία θα καταλήξουμε σε συμφωνίες για τα έσοδα χωρίς να συμβάλλουμε στην ε, διαρκή δημιουργία δορυφορικών μέσων προς τον προϋπολογισμό, οι οποίοι θα απομακρύνουν τελικά από την κεντρική διοίκηση. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ανάγκη και θα πρέπει να συμφωνήσουμε γι' αυτό. Θα γίνει και μια συνάντηση των σκιωδών, θα συζητήσουμε διάφορα στοιχεία. Θα δούμε τι θα γίνει και με το δεύτερο ημίση των παραγράφων της έκθεσης. Νομίζω ότι σίγουρα χρειαζόμαστε του EFSM, ε, αλλά θα πρέπει να δούμε και στο μέλλον τι θα γίνει, γιατί στο μέλλον θα έχουμε 27 κρατημέλη, εκ των οποίων ένα έχει επιλέξει ρητά το opt-out και οι υπόλοιπε ε, χώρες εφόσον ε, το επιθυμούν και εφόσον είναι έτοιμες, μπορούν να ενταχθούν στη ζώνη ευρώ. Και έτσι λοιπόν διαμορφώνεται μια νέα κατάσταση και θα πρέπει όλα να λεφθούν υπόψη για να αποφευθούν παράλληλες δομές. και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι χώρε αυτέ να ενταχθούν ενδεχομένω στην Ευρωζώνη και να παραμείνουν παρούσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρο, και πρωτού ολοκληρώσουμε, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ θα λάβει χώρα το Σεπτέμβριο. Η στις 26 ε, Σεπτεμβρίου και στην Ολομέλεια κατά την δεύτερη Ολομέλεια του Οκτωβρίου.